Έχουμε μια σύντομη παρουσίαση τη έκθεση Νίνα Γκίλ για την αποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μα. Δεν σα είχα δει, με συγχωρείτε, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πίσω από αυτή την έκθεση για την διαβούλευση ω πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ανησυχία ότι καθυστερημένη πληρωμή οφειλών είναι εις βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά την έλλειψη πληροφοριών σε σχέση με τους ε, οφειλέτες και εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι όταν βρίσκεται σε σχέση με τον οφιλέτη, όταν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι δυνατόν να ανοιχνευτεί ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Και εδώ σε σχέση με τις διατάξεις σας, σε σχέση με τα εθνικά νομικά πλαίσια, να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε μητρό πληθυσμού. Εδώ Τίθενται ερωτήματα αν ε, οι αρχές ε, δίωξης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους ε, στοιχεία καθώς επίσης και σε φορολογικά μητρώα καθώς επίσης σε σχέση με την βελτίωση πρόσβασης σε αυτά τα στοιχεία των φορέων για την δυνατότητα υποχρέωσης των χρεωστών να αποκαλύπτουν μέσα στο ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο όλα τα στοιχεία τους και σε σχέση με την έκθεση μου, η ε, θα υπήρχε όφελος από την εισαγωγή ενιαίων πιο ευέλικτων διαδικασιών που θα εφαρμοζόντουσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί εντολή για την αποκάλυψη τέτοιου είδους και γνωστοποίηση τέτοιου είδους στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε ε, δικαστική απόφαση. Δίνεται η δυνατότητα έτσι άμεσης ε, πληρωμής ε, ή άμεσης εξόφλησης. Η έκθεση επίσης ζητεί να υπάρξει μία μελέτη ώστε να μπορούν να υπάρχουν δυνατότητες σύγκρισης σε σχέση με την εφαρμογή με χώρες παραδοσιακού εθνικού δικαίου common law όπως τη Μεγάλη Βρετανία και ευρωπαϊκές χώρες ε, ε, στις οποίες ισχύει το ρωμαϊκό δίκαιο και την δυνατότητα να μπορεί να διασφαλίζεται και το θέμα των ε, προσωπικών στοιχείων αλλά και να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου. Πρέπει να γίνει αυτό ώστε να είναι δυνατόν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των νομικών συστημάτων κρατών μελών να αντιμετωπιστούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πολλές από τις προτάσεις μας θέλουν την πρόταση να την κάνουν πιο διαφανή και να είναι πιο ευέλικτη η διαδικασία. Γι' αυτό είναι σημαντικό το ε, εγχειρίδιο της ε, ε, εφαρμογής των πρακτικών να επικαιροποιείται και οι πληροφορίες να διατίθενται σε ένα, με, σε τρόπο, που θα είναι εύκολο να χρησιμοποιούνται. Κέρια σημασία είναι να μπορούμε να δραστηριοποιούμαστε ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε παράλληλα το έργο των εθνικών αρχών και όχι να υποκαθιστούμε τις δράσεις αυτές λαμβάνοντας πάντα υπόψη πόσο σημαντικό θα είναι να μπορεί να λειτουργεί αυτή η νομοθεσία αποτελεσματικά. Έτσι θα μπορέσουν να ε, ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να βοηθηθούν να ξεπεράσουν ένα σημαντικό πρόσκομα διότι δεν έχουν ε, τους πόρους ε, όπως έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις να ε, προβούν σε διώξεις εις βάρος οφειλετών που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Και αν λοιπόν αποθαρρύνονται οι επιχειρήσεις λόγω προσκομμάτων, αυτό δημιουργεί απειλή για την σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει να είναι θεμελιώδου σημασία να διασφαλίζουμε τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιχειρήσεις έχουν ένα μεγάλο ε, ποσοστό των επιχειρήσεών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω για την ε, υποστήριξη που μου δόθηκε στη σύνταξη αυτής της έκθεσης και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους άλλων ομάδων για την επικοδομητική αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Αυτό το οποίο έχει σπουδαιότητα σε αυτή την νομοθεσία που θέλουμε να προαχθεί είναι το ότι θα πρέπει να ακολουθήσει κατεπηγόντως ε, το έργο αυτό και τις προτάσεις της Ευρωβουλής η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεγάλο μέρος ε, θα πρέπει να επικεντρώνεται σε πραγματικά ε, τις ε, σωστές διαστάσεις των επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ Κύριο Επίτροπος έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε δυνατότητα να συζητήσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα τη διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέ. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν συμφωνήσει για την διασυνορική ανάκτηση των ε, οφειλόμενων ποσών και θεωρούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και η προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά των οφειλετών αυτών. Επίσης είπαμε ότι είναι σημαντικό για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στην σημερινή ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Οι αρχές ε, τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα θα πρέπει να διέπουν και του στόχους της κοινότητα που διαθέτει μια πάρα πολύ εντυπωσιακή δέσμη νομικών μέτρων για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας και παρόλα αυτά σίγουρα το πρόγραμμα βίας αναγνώρισης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δείχνει ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο να υπάρχει επιβολή των αποφάσεων, των δικαστικών αποφάσεων ε, στο έδαφος ε, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Και υπάρχει και η πράσινη βίβλος του 2008 όλες οι απαντήσεις ε, και η σύνοψη μπορούν να μελετηθούν από τους ενδιαφερόμενους στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Και μάλιστα ε, υπάρχουν και συγκεκριμένες απόψεις για το τι μπορεί να γίνεται στην πράξη για την επίλυση των προβλημάτων. Η έκθεση της κυρίας ε, Τζιλ εκφράζει κάποια δυσπιστία σε κάποιες ε, απόψεις, θεωρώντας ότι το βασικό πρόβλημα είναι οι υποτροπιάζοντες, ας πούμε, οφειλέτες. Και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνονται κάποια στοιχεία για την οικονομική κατάσταση ορισμένων ατόμων. Θα πρέπει να δούμε όμως και το θέμα των, προσωπικού, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να δούμε επίσης αλλοδαπούς οφειλέτες που εργάζονται σε άλλα κρατημέλη θα πρέπει να δούμε τι προσωρινά μέτρα μπορούν να ληφθούν. Η βελτίωση της πρακτικής εφαρμογής των ε, δικαστικών αποφάσεων θα αποτελέσει προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο ε, του προγράμματος της Στοκχόλμης για την περίοδο 2010-2014. Τον Ιούνιο του 2009 θα υποβάλει το πρόγραμμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια δεν έχουμε ακόμη προγραμματίσει κάποια συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα ως ε, συνέχεια σε αυτό το πράσινο βιβλίο. Τέλος, και υπό το πρίσμα των πρώτων αποτελεσμάτων ε, της διαβούλευσης που είχαμε πιστεύουμε ότι η πρόταση για την αύξηση της πρόσβασης ε, στα δημόσια μητρώα, για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, και για την δημιουργία μιας ε, υπεύθυνη δήλωσης από τον Φιλέτη πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση την εκπλήρωση των στόχων μας, αλλά θα πρέπει σίγουρα να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα διάφορα θέματα τα οποία περιλαμβάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 12 στη συνέχεια μου την παρουσίαση της κυρίας Μαγκίνες για ε, την ετήσια έκθεση για τις διαβουλεύσεις Επιτροπής Αναφορών 2008. Το λόγο στην εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι.